Is that that's on now? If colleagues could take their seats, then we could. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε γρήγορα.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 Ίσως γιατί είμαι το παλαιότερο μέλος του Κοινοβουλίου ενώ σε αυτή την Επιτροπή. Σας καλωσορίζω όλους και τα παλαιά μέλη που επανήλθαν και τα νέα μέλη. Στόχος μας σήμερα είναι μόνο να συνθέσουμε το Προεδρείο δηλαδή τον πρόεδρο και τους τέσσερις αντιπροέδρους επί τη βάση του άρθρου 113. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε το 213 η σειρά της εκλογής είναι πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο και μόλις εκλεγεί ο νέος πρόεδρος θα πάρει τη θέση μου και θα συνεχίσει την διαδικασία για την εκλογή των τεσσάρων αντιπροέδρων. Πρώτος μου στόχος, αποστολή μάλλον, είναι να πω ότι ορισμένα μέλη <laughs> Substitutes. So Mr. Pizarro will replace Mr. Bradford for Λοιπόν, θα αντικατασταθεί ο κύριος Μπράτφορτ, για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Ράισεν θα αντικαταστήσει τον κύριο Τόμασεκ από το ECR και η κυρία Χάζεμπκάμπ θα αντικαταστήσει τον κύριο Φερέρα για την ΚΟΕ. Και ίσως να υπάρχει και άλλη μία αντικατάσταση. Θα ήθελα να πω ότι το Ευρω... η σοσιαλιστική ομάδα έχουμε άλλον ένα αναπληρωτή στη θέση του κυρίου Μπαρτόλο αντικαθίσταται από τον κύριο Γκονσάλες Κατσάρες. Θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπαρτόλο. Έχουμε δηλαδή συνολικά δύο αναπληρωτές εμείς. Καλώς. Υπάρχει κάποιος άλλος. Ο Μάνερη που είναι αναπληρωτής θα αντικαταστήσει την Dodge. Η Τζούν είναι εδώ μαζί μου. Είναι για τους μη εγγεγραμμένους. Εντάξει. Καλώς αν δεν υπάρχουν άλλοι αντικαταστάτες. Ε, θα πρέπει να ελέγξουμε την απαρτία. Είναι σαφές ότι υπάρχει απαρτία. Χρειαζόμαστε το 25% ε, και υπάρχει. Τώρα, ε, θα ήθελα να ζητήσω τις προτάσεις για την εκλογή. Το Renew Europe προτείνει την υποψηφιότητα του κυρίου Chris Davis για την Προεδρία της Αλίας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη πρόταση για τη θέση του Προέδρου. Δεν υπάρχουν ε, άλλες προτάσεις. Τότε θα ζητήσω από τον υποψήφιο αν δέχεται την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δέχομαι για την πρόταση φαίνεται να υπάρχει μόνο μία πρόταση, οπότε έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε διαβοής, εκτός αν το 1 πέμπτο των μελών, δηλαδή 6 μέλη, ζητήσουν μυστική ψηφοφορία. Αν δεν έχει αιτηθεί κάποιος μυστική ψηφοφορία, τότε μπορούμε να ανακηρύξουμε ε, τον κύριο Ντέιβις, πρόεδρο της Επιτροπής μας.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 Um, Καλώς συνάδελφοι, είμαστε η μικρότερη επιτροπή, αλλά στη μεγαλύτερη αίθουσα. Δεν θα ξαναδούμε τόσο μεγάλες αίθουσε. Υπάρχουν πολλά νέα μέλη. Εδώ είναι ο κ. Κουάντε, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της γραμματείας. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα στη γραμματεία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, ποιος μάλλον διαχειρίζεται τα πράγματα στην Επιτροπή μας. Σύντομα θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή αυτή τα τελευταία χρόνια έχει κάνει καλή δουλειά, έχει βοηθήσει την βιωσιμότητα των αλλιευμάτων σε πάρα πολλές θάλασσες, υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, ελπίζω τα επόμενα χρόνια ε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε η αλλιευτική δραστηριότητα να αναπτυχθεί. Θα ήθελα να περάσω στο επόμενο θέμα λοιπόν που είναι η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Ποιος ε, προτείνει ποιον. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προτείνω τον κύριο Βαντάλεν, Πίτερ Βαντάλεν. Πρώτος αντιπρόεδρος. Δέχεστε την πρόταση, ναι λέει ο κ. Βαντάλεν. Υπάρχουν άλλες προτάσεις, όχι. Συνεπώς διαβοής γίνεται δεκτή η πρόταση, ο κ. Βαντάλεν είναι αντιπρόεδρος. Fabio. Um, I think it, it is probably apposite that I point out, as we now have a male. Έχουμε άντρες πρόεδρο και αντιπρόεδρο, πρέπει να πω, οπότε καλό θα ήταν να διαφοροποιήσουμε λιγάκι εδώ τα, τους συμμετέχοντες στο Προεδρείο να δούμε πώς θα είναι οι επόμενες ψηφιότητες. Δεύτερος αντιπρόεδρος. Η ομάδα Renew Europe σας προτείνει με χαρά την υποψηφιότητα του Σορέν Γκαντζό. Συμφωνείτε? Ναι κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Άλλη για δεύτερη αντιπροεδρία, πάλι διαβόηση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 Thank you. I seek nominations for the position of third. Πάμε στον τρίτο αντιπρόεδρο. Έχετε υποψηφιότητες να υποβάλλετε. Παρακαλώ. Η κυρία Κλάρα Αγγιλέρα. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, κύριε Ντέιβις, και να στείλω και ένα μήνυμα στο Βρετανικό λαό. Εμείς αγαπούμε πολύ τους Βρετανούς να δούμε αν εκείνοι αγαπούν την Ευρώπη. Το, εσείς το ξέρω. Ε, θέλω να είναι ένα θετικό μήνυμα προς το Βρετανικό λαό. Βγάλαμε πρόεδρο Βρετανό στην Επιτροπή Αλίας. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι η σοσιαλιστική ομάδα καταθέτει την υποψηφιότητα του κυρίου Τζουζέπε Φεραντίνο για ε, τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Είναι γεγονό ότι είμαι Βρετανός. Ε, Αναφανδών υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν χάνω ευκαιρία ε, να πείσω ε, τη χώρα μου να παραμείνουμε και να μην αποχωρήσουμε στις 31 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. So we have received a nomination Λοιπόν, λάβαμε υποψηφιότητα για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Δέχεστε, βεβαίως. Ναι. Άλλες υποψηφιότητες.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 Σα θυμίζω <laughs> την ισορροπία του φίλου για την τέταρτη θέση αντιπροέδρου. Έχουμε υποψηφιότητε. Παρακαλώ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά και τιμή σα υποβάλλω την υποψηφιότητα της κυρία Σοζάνα Κόντε που θα βάλει και ε, την εκπροσώπηση του γυναικείου φίλου πέρα από τις ικανότητές της φυσικά στο Προεδρείο της Επιτροπής αυτή. Κυρία Κόντε, δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Ναι, τι δέχομαι, ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες. Ο κύριος Μιγιάν Μον. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να καταθέσω την υποψηφιότητα της κυρίας Κλάουδια Μοντέρο ως τέταρτη αντιπρόεδρο. Συμφωνείτε, δεν το δέχεστε, ναι. Ωραία, άρα έχουμε δύο υποψηφίους και θα πρέπει να ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία. Χρειάζεστε τις κάρτες σας. Θέλετε εξηγήσει για το πώς λειτουργούν τα μηχανήματα. Πάει καιρός που δεν έχω χρησιμοποιήσει εγώ τέτοιο μηχάνημα, μια πενταετία. Right. So um, um, Λοιπόν, έχουμε δύο υποψηφίους. Για να ψηφίσετε θα πατήσετε το πράσινο ε, κουμπί για την κυρία ε, Κόντε και το κόκκινο για την κυρία Μοντέρο. Εντάξει. Το πράσινο κουμπί είναι για την κυρία Κόντε. Το κόκκινο για την κυρία Μοντέρο. vote is open. Έρχεται η ψηφοφορία. Has everyone voted? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επομένως, εκλέγεται κυρία Μοντέρο. Please take the plate.